Καλησπέρα σας, παρακαλώ, καθίστε. Καλωσορίζω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους των Εθνικών Αντιπροσωπείων των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή την συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω θερμότατα και ιδιαίτερα εγκάρδιο χαιρετισμό απευθύνω στη συμπρόεδρό μου, την κυρία Ταλβιτή, που εκπροσωπεί τη Φιλανδική Προεδρία, την εκπεριτροπή δηλαδή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φιλανδία, όπω ξέρετε, ασκεί την Προεδρία στο τρέχον εξάμεινο. Οπότε θα έχουμε συμπροεδρία στη σημερινή συνεδρίαση. Θα ασκήσουμε την Προεδρία από κοινού η ε, κυρία Ταλβίτη και ο υποφαινόμενο. Χαίρομαι μεγάλη χαρά και τιμή που σα υποδέχομαι εδώ σε αυτή την πέμπτη συνεδρίαση Τη μεικτή ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, GPSG όπω τη λέμε. Πολύ σημαντική ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου για τη Europol. Την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία σε θέματα ασφάλεια δηλαδή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που 64 εθνικά κοινοβούλια εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Διορθώνει ο πρόεδρος. 64 ε, βουλευτές από εθνικά κοινοβούλια, από 36 κοινοβουλευτικά σώματα και 26 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα και το υπαριθμό ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης. είχαμε αρκετή πρόοδο από τελευταία δεκαετία με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το και τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπλήρωσε τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ενίσχυσε το ρόλο τη Ευρωπόλ στα θέματα τη αστυνομική συνεργασία. Οι αστυνομικέ αρχέ και άλλε υπηρεσίε ε, επιβολή του νόμου έχουν αμοιβαία συνεργασία προκειμένου να προλάβουν και να καταπολεμήσουν, σοβαρό έγκλημα διασυνοριακού χαρακτήρα δύο και κρατών μελών και φυσικά να αντιμετωπίσουν ε, εγκλήματα του κοινού ποινικού εφόσον βάλλονται κατά το κοινωτικών συμφερόντων. Και εμεί, η μεικτή αυτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, ασκούμε ακριβώ τον, όπω λέει και το όνομα, ο τίτλο τη ομάδα μα, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ευρωπόλ. Και με σε στενή συνεργασία, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται και διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο της Ευρωπόλ. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα... Το πρόγραμμα μας είναι ιδιαίτερα έντονο, γι' αυτό και σας θέλω παρακαλώ να έχετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα και την στενότητα χρόνου. Σήμερα έχουμε δύο συνόδους και αύριο το ίδιο. Ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο τμήμα, μετά την πρώτη σύνοδο θα έχουμε ένα διάλειμμα για καφέ, θα έχουμε δεύτερο, δεύτερη σύνοδο και μία τρίτη φάση όπου θα έχουμε ε, καλεσμένο τον κύριο Πελεγκρίνη και τον αναπληρωτή επόπτη προστασίας δεδομένων. Βέβαια, προβλέπουμε χρόνο και για συζήτηση, όπως πάντα, σε διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Και εδώ έχουμε προβλέψει χρόνο για συζήτηση. Και θα δίνω εκ περιτροπής το λόγο σε εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές. Αλλά θέρμο παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, κατάμεστη σε διάταξη. Και μόνο αν τηρούμε το χρόνο αγόρευση θα καταφέρουμε να τη διεκπαιρεώσουμε ε, έγκαιρα. Όπως σας είπα, σήμερα θα έχουμε να κάνω δύο γύρους συζήτηση στους αρχικούς και θα ακούσουμε την προστασία, την παρουσίαση από τον αναπληρωτή επόπτη προστασία δεδομένων, τον κύριο Βιεβουρόφσκι. Θα ξεκινήσουμε όμως με την εκτελεστική διευθύντρια της Europol, που βρίσκεται εδώ στο Προεδρείο. Καλώς ήρθατε κυρία Ντεμπόλ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ. Έχουμε και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ, τον κύριο Λίντσα, Αντρέι Λίντσα. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Σήμερα το βράδυ, κεντρικός ομιλητής της διάσκεψής μας θα είναι ο Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας, που βρίσκεται στο τελευταίο τμήμα της κοινοβουλευτικής του, της θητείας του, της πενταετούς θητείας του, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά τις ε, συνόδους που θα έχουμε, θα παραθέσουμε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεξίωση. Θα έχουμε λοιπόν και εκεί κάποιο χρόνο για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Πάντως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες τροπολογίες που αφορούν τη συμμετοχή της Δανίας στη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε από τους συμπροέδρους μετά την πρόταση στην ομάδα εργασία για τη συμμετοχή της Δανίας. Και οι συμπρόεδροι και η τριάδα της Προεδρίας ε, πρότειναν τη συμμετοχή της Ισθανία. Και μάλιστα σήμερα έγινε μια παρασκευαστική συνεδρίαση της Τριάδας των Προεδριών και κατά εξαίρεση ε, καλέσαμε την γερμανική αντιπροσωπεία ως συνομιλητή σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης. Γιατί η γερμανική προεδρία θα ακολουθήσει την Κροατική Προεδρία. Η Ρουμανία, η Φιλανδία και η Κροατία συνιστούν την τριάδα των Προεδριών. Η κυρία Τελβιτιέ είναι εκπρόσωπος της Φιλανδικής Προεδρίας, της τρέχουσας και θα μας ενημερώσει για τη σχετική συνεδρία. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να καλωσορίσω και επισήμως την κυρία Μέριλίνα Τελβιτιέ που είναι επικεφαλής της Φιλανδικής Αντιπροσωπείας ε, στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτήν την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές ε, και κύριοι βουλευτές αγαπητοί προσκεκλημένοι. Σας ε, καλωσορίζω πρώτα απ' όλα και μεγάλη μου χαρά το ότι ε, συναντώμαστε για πέμπτη φορά είναι κάτι το οποίο οργανώνουμε από κοινού με το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όταν ιδρύθηκε η Europol. Αυτό είναι κατόπιν απέτησης των κρατών για να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή εγκληματικότητα. Ο κανονισμός της Europol ετέθη πριν από ισχύ, πριν από ετέθη ενισχύ πριν από αρκετά χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια ενίσχυση των εθνικών διοκτικών αρχών και ε, διάφορων άλλων μονάδων, ε, ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Ε, ταυτόχρονα υπάρχουν εκπαιδευτικές αρμοδιότητες της Europol, στόχος των οποίων είναι η επίτευξη καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Europol και κρατών μελών, πάντα βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της ε, Europol ε, και η ανταλλαγή πληροφοριών με τα κοινοβούλια θεωρήθηκε ιδιαίτερο σημαντικός, γι' αυτό έχουμε τακτικά τις ε, σχετικές συνεδριάσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα και αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται ακριβώς στο ότι έχουμε κάποιες κοινέ αξίες, στο ότι είμαστε ενωμένοι. Είναι λοιπόν για μια χώρα μόνη της αδύνατον ε, να καταπολεμήσει το διεθνές έγκλημα και την τρομοκρατία. Μόνο από κοινού μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Europol λοιπόν προσφέρει στα εθνικά κράτη γνώση ε, δυνατότητες, ε, πληροφορίες ε, για να κάνουν κάποια πράγματα που δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν μόνα τους ή δεν θα είχαν τους πόρους. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό η Europol να έχει επαρκείς πόρους για να ανταποκριθεί στην αποστολή της Έχουμε συνεργασία ακριβώ για να καταπολεμηθούν τα σοβαρά εγκλήματα και αυτό είναι σημαντικό ανεξαρτήτως του σε ποιο κράτος ζει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχηθώ μια καλή συνεργασία, έναν καλό διάλογο ε, και κατόπιν θα συνεχίσω στα αγγλικά. um... Θα ήθελα να σας ενημερίσω επίσης για την συνάντηση της Προεδρικής Τρόικα, της Τρόικα της Προεδρίας, που έγινε σήμερα το πρωί. Συζητήσαμε τα εξής. Το σχέδιο μερίσιας διάταξης της ε, μικτής κοινοβουλευτικής διάσκεψης, τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας για τη συμμετοχή της Δανίας, το θέμα του ορισμού εκπροσώπου της Μεκτής Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης ε, που θα πάει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, ε, τροποποιήσεις του κανονισμού και γραπτές παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Επίσης έγινε ανταλλαγή απόψεων με τον επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής καθώς η, Γερμανία θα αποτελέσει μέλος της Τρόικας από το επόμενο εξάμεινο. Ο κανονισμός προβλέπει την ε, δυνατότητα οι βουλευτές να αποστείλουν γραπτές ε, ή να απευθύνουν προφορικές ερωτήσεις ε, προς την Europol. Οι συμπρόεδροι έχουν λάβει από την τελευταία συνεδρίαση μια ερώτηση από ε, μια βουλευτή και είχε προβλεφθεί μια διορία για την απάντηση 6 εβδομάδων. Λάβαμε την απάντηση την Παρασκευή και την μοιράσαμε στους βουλευτές. Επιπλέον, από την τελευταία μας συνεδρίαση κάποιες ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την προηγούμενη συνεδρίασή μας έχουν εντωμεταξύ απαντηθεί από την Europol και προωθήθηκαν οι απαντήσεις αναλόγως. Έχουμε τώρα την έγκριση της μερίσιας διάταξης της πέμπτης μικτής κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε όλοι λάβει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης από την Τρόικα της Προεδρίας. Έχετε κάποια σχόλια? Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Η έναρξη της Ολομέλειας. Ας ξεκινήσουμε τώρα την Ολομέλεια. Τη πέμπτη της ε, συνεδριασής μας. Περνάμε στο πέμπτο σημείο της ημερήσια διάταξη. Αναφορά δραστηριοτήτων της Europol από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο του 2019 και σχεδιο πολιετου πολιτού προγράμματος 2020-2022. Πριν ε, ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της κοινότητας, ε, εκτός ε, από την Ιρλανδική. Παρακαλώ δείτε τις οδηγίες ε, που υπάρχουν μπροστά σας. Εκεί θα δείτε και πώς θα συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Η διάσκεψή μας μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και σας εύχομαι παραγωγική εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Συμπρόεδρε, κυρία Ταλβίτη, περνάμε τώρα στα ουσιαστικά ζητήματα του ημεσίου, της ημερησίας διάταξης όμως απασχολήσουν για δύο μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν με την παρουσίαση που θα μας κάνει ο ή ε, κύρια ομιλητή μα, η κυρία Κάθριν Ντεμπόλ, εκτελεστική διευθύντρια τη Europol, η οποία θα μα παρουσιάσει δραστηριότητε από τον Μάρτιο 2019 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2019, τις κύριες προκλήσεις ε, μεταξύ των οποίων και ο προπολογισμό και τις προοπτικές. Όλα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού περί Europol για το σχεδιο πολυετους πολιετούς προγράμματος 2020-2022. Στρατηγική αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο η Europol να αποτελέσει έναν κόμβο για ε, ζητήματα εγκληματικότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε ήδη μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην συνάντησή μας στο Βουκουρέστι τον Φεβρουάριο. Τώρα, δύο λόγια για την οργάνωση της συζήτησης. Όσοι γνωρίζετε τις ε, διακοινοβουλευτικές διασκέψεις θα γνωρίζετε πως ε, οργανώνουμε κύκλους ερωτήσεων και απαντήσεων και σε κάθε τέτοιο κύκλο θα έχουμε δύο βουλευτές Εθνικών Κοινοβουλίων που θα λαμβάνουν το λόγο. Ναι, και έναν Ευρωβουλευτή. Εάν θέλετε λοιπόν να λάβετε τον λόγο, σας παρακαλώ, ε, στείλτε εδώ στην γραμματεία τα έντυπα που έχετε μπροστά σας ε, ή θα σας τα μοιράσουν συμπληρώστε το όνομά σας, ε, την ιδιότητά σας και θα σας δώσουν χρόνο ομιλίας. Όπως είπα, δύο εθνικοί βουλευτές ε, και ένας ευρωβουλευτής σε κάθε γύρο. Για να ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ημερήσια διάταξη, την απόψινή και την αυριανή. Οπότε ε, σας παρακαλώ να είστε λογικοί στον χρόνο ομιλίας. Ε, προτείνω λοιπόν να περιοριστεί ο καθομιλητής στα δύο λεπτά. Έτσι ώστε και ο Προεδρεύων να έχει τον χρόνο και ο μιλητής βεβαίως, στον οποίο απευθύνεται τις ερωτήσεις, να μπορέσει να απαντήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας βοηθήσετε και εσείς στην διεξαγωγή. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της κυρίας Ντεμπολ, εκτελεστικής ε, διευθυντρίας της Europol. Σας ε, καλωσορίζω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε τον λόγο για τα επόμενα 15 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγελάρα, κυρία Μαριλένα Τελβίτη, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στην μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου για την Ευρωπόλ. Θα ήθελα να σας αναφέρω τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το πολιετές προγραμματικό έγγραφο ε, μέχρι το 2022 της Ευρωπόλ καθώς και τις γραπτές ε, ε, συνεισφορές που έχουμε λάβει μέχρι, τότε και θα, μέχρι σήμερα και θα σας δώσω και κάποιες επιχειρησιακές, κάποια επιχειρησιακή ενημέρωση από την τελευταία συνεδρία στο Βουκουρέστι για το πολιετές έγγραφο 2022. Θα θυμάστε στην τελευταία συνάντηση σας έδωσα μια γενική επισκόπηση. Παρουσίασα την στρατηγική της Ευρωπόλ, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Σύμβουλο της Ευρωπόλ, αποτελούμενο από μέλη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η στρατηγική 2020 Plus αποτελεί τη βάση για το πολιετές προγραμματικό έγγραφο της Ευρωπόλ. Δράτω τη ευκαιρία για να σα επισημάνω τα βασικότερα στρατηγικά στοιχεία του εγγράφου αυτού και να σα ενημερώσω για τι τελευταίε εξελίξει που σχετίζονται με την υλοποίηση τη στρατηγική τη Ευρωπόλ. Οι ακόλουθε προτεραιότητε είναι οι εξή. Πρώτη, η Ευρωπόλ θα αξιοποιήσει στο έπακρο τι πληροφορίε που λαμβάνει από ένα εκτενέ δίκτυο εταίρων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, θέλουμε να είμαστε ε, ο κόμβος ε, ποινικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε απλά να συλλέγουμε δεδομένα, αλλά και να διασυνδέουμε τις πληροφορίες. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι λοιπόν περισσότερο από παλιά ε, και να υποστηρίζουμε επιχειρησιακά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα εστιαστούμε στις υποθέσεις προτεραιότητας, τις έρευνες που έχουν προτεραιότητα για προ στόχου υψηλή, αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να κυνηγήσουμε του πιο εξελιγμένου και επικίνδυνου εγκληματίε με την υποστήριξη πολυτομιακών ομάδων. Τρίτον, η Ευρωπόλ πρέπει να γίνει πλατφόρμα για τι ευρωπαϊκέ ε, λύσει αστυνόμευση. Και τέταρτον, θα πρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή τη καινοτομία και τη έρευνα ε, στον τομέα τη επιβολή του νόμου. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να γίνει ένα οργανισμό καινοτομία και φορέας καινοτομέ. Η υλοποίηση τη στρατηγικη 2020+ σε επιχειρησιακούς όρους μεταφράζεται σε ισχυρή εστίαση στους ε, ε, βασικούς στόχους προτεραιότητας. Αυτή είναι η βασική απασχόληση των αστυνομικών αρχών. Το 2019 έχουμε κάνει και επιχειρησιακές προσαρμογές που θα δημιουργήσουν συνέργειες και θα μας βοηθήσουν να εστιαστούμε στου πόρους σε τομεί προτεραιότητας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε συστήσει μια task force ανάλυσης, μια task force αρμόδια για την δημιουργία του νέου κέντρου χρηματοοικονομικού και οικονομικού κλίματος, ένα έργο καινοτομίας και το ε, προγραμματικό συμβούλιο διαχείριση πληροφοριών. Η Task Force Ανάλυσης θα εργάζεται για την ενίσχυση της δικής μας ανάλυσης και των αναλυτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε μια online ε, πλατφόρμα ανάλυσης. Έχουμε λάβει ε, μια ενθουσιώδη απόκριση από πάνω από 800 αναλυτές ε, από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να μοιραστούν μαζί μας γνώση, εμπειρογνωμοσύνη και εργαλεία. Όπω είπα η Task Force ε, για το νέο κέντρο χρηματοοικονομικού και οικονομικού εγκλήματο. θα σχεδιάσει το νέο κέντρο, θα καθορίσει τη δομή και τι απαιτήσει του κέντρου προ υποστήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού και οικονομικού εγκλήματο, συμπεριλαμβανομένης τη διαφθοράς. Το ε, Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείριση Πληροφοριών θα καθορίσει το κοινό όραμα και το αντικείμενο τη ε, διαχείριση πληροφοριών στην Ευρωπόλ. Το έργο καινοτομία θα εστιαστεί στη χαρτογράφηση του τοπίου καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την άποψη τη επιβολή του νόμου. Θα βοηθήσει να αναπτυχθεί μια στρατηγική καινοτομία και μια δομή διακυβέρνηση τη καινοτομία που θα βοηθήσει οι πληροφορίε να αποτελούν απόσπαστο κομμάτι στο μέλλον. Αυτή είναι η τομή των νέων εξελίξεων που σχετίζονται με το πολιετέ προγραμματικό έγγραφο 2020. Παράλληλα με αυτό, θα ενισχύσουμε επιπλέον περαιτέρω ε, τρία ε, ήδη υπάρχοντα επιχειρησιακά κέντρα στην Ευρωπολ, ε, το, για το κυβερνοέγκλημα, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το κέντρο σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Για παράδειγμα, η Ευρωπόλ θα ήθελε να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, την κατάλυση τρομοκρατικού περιεχομένου online και την διάσωση παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάχρηση όπως είπα νωρίτερα. Πρόκειται για μια στρατηγική για μετά το 2020. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Ωστόσο, οι επενδύσει στην Ευρωπόλ είναι επενδύσει απευθεία στην υποστήριξη των αρχών επιβολή του νόμου των κρατών μελών. Αυτή η τελευταία παρατήρηση με οδηγεί στο νέο θέμα επαρκής χρηματοοικονομικές και, ε, χρηματοοικονομική και ανθρώπινη πόρη για τον οργανισμό μας. Κάτι ζωτικό για να μπορούμε να παράσχουμε την προστιθέμενη αξία και βελτιωμένες υπηρεσίες. Η Ευρωπόλ χρειάζεται έναν βιώσιμο προπολογισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση μακροχρόνιων επενδύσεων που θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μας επιχειρήσεις. Η συνολική κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχει με στόχο, με γνώμονα την ανάπτυξη. Όχι για, απλά για να υπάρχει, για να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση, την αυξανόμενη ε, κοινότητα χρηστών, ε, μια, ένα ε, ευρύτερο αντικείμενο και μια ευρύτερη εντολή, τι σοβαρές απειλές στην ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την JPSG για την υποστήριξή της κατά τις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού 2020 και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Καλωσορίζω την γνωμοδότησή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τον προπολογισμό 2020 που υποστηρίζει πλήρως το, τα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ για το 2020. Ο Περσεμένη 173,6 εκατομμύρια ευρώ και 66 επιπλέον μέλη του προσωπικού. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κρατημέρη να μπορέσουν να ακυρώσουν αυτή τη θέση. Ακόμη και αν η τελική έκβαση του προπολογισμού ε, παρότι δεν είναι ακόμα γνωστή η τελική έκβαση, η μορφή του προπολογισμού, η βοήθεια σα δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό όραμα για το τι στήριξη θα πρέπει να λαμβάνει και να παρέχει η Ευρωπόλ στα κράτη-μέλη. Το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθορίσει τα ανώτατα όρια των πόρων μα για την περίοδο 2021-2027. Η σημερινή πρόταση προβλέπει σοβαρέ περικοπέ στον προπολογισμό τη Ευρωπόλη. Για παράδειγμα, εκτιμάται σήμερα περικοπή άνω του 10% για το 2021 στον προπολογισμό τη Ευρωπόλ σε σχέση με τον σημερινό προπολογισμό τη. Πλησιάζουμε τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με μια συμφωνία που θα γίνει ε, δεκτή στα τέλη του έτους. Ελπίζω οι εθνικές κυβερνήσεις να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ευθυγράμμιση του προπολογισμού της Ευρωπόλ με τις επιχειρησιακές και πολιτικές απαιτήσει. Θα ήθελα να απαντήσω στις γραπτές ε, συνεισφορές στο προγραμματικό έγγραφο της Ευρωπόλ 2022 που λάβαμε από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία, την οποία ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα σχόλια. Η Ευρωπόλ αυτή τη στιγμή ε, στέλνει δύο με τρεις ε, ε, αξιωματικούς στην Κύπρο. Από τις 3 Απριλίου του 2019 υποστήριζε τις αρχές επιβολής του νόμου της Κύπρου η Ευρωπόλ στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου για δευτερεύοντες ελέγχους ασφαλείας στην Κύπρο. Προσκεκλημένοι αξιωματούχοι της Ευρωπόλ λειτουργούν σε ένα γραφείο στο ε, τμήμα μετανάστευσης μπορούν να κινούνται στη Δημοκρατία της Κύπρου όπως απαιτείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ, των αξιωματούχων της και όλων των αρμόδιων αρχών έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και υπάρχει μια υγιής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, Κυπριακών Αρχών και της Ευρωπόλ. Όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση και τα κρυπτονομίσματα αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να συμφωνήσουμε για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ε, κρυπτογράφησης μαζί με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η Ευρωπόλ προσπαθεί να προχωρήσει τις, ε, την στρατηγική της αυτό το τομέα ε, στο πλαίσιο των πόρων που διαθέτει. Αποτελεί ζήτημα κλειδί για ολόκληρη την κοινότητα επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες, θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση για τους ακόλουθους τομείς ε, εγκλημάτων, κυβερνοέγκλημα, η δομή των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ξέπλυμα μαύρου χρήματο και παιδική πορνογραφία. Στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος αυτή τη στιγμή τα ransomware είναι η πρώτη απειλή που αναφέρεται στον τομέα των κυβερνοεπιθέσεων. Με στόχο πολίτες, ε, ε, με στοχευμένες εκστρατείες κατά επιχειρήσεων ζητώντας ε, λίτρα έως και ε, εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε σχετίζεται με το ransomware Goga όπου ε, γίνεται επίθεση σε βιομηχανικές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Εμείς δημιουργήσαμε μια ομάδα, ένα κέντρο αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος και μια task force για την καταπολέμηση αυτής της συγκεκριμένης οικογένειας λιτρισμικών. Ε, μια άλλη δυσκολία είναι το σκοτεινό δίκτυο. Η συντονισμένη δράση του Cyber Crime Center ε, συγκεντρώνει διάφορους εθνικούς εμπειρογνώμονες για τον εντοπισμό των στόχων στο Dark Web από 273 στόχους που είχαν ε, καταρτιστεί αρχικά σε ένα κατάλογο. 206 ε, αντιμετώπισε βασικά η Ευρωπόλ και οι τρεις βασικοί κλάδοι είναι τα πυροβόλα όπλα, το κυβερνοέγκλημα και τα ναρκωτικά. Το, οργανωτικό έγκλημα στην Ευρωπαϊκή, το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Οι βασικές ομάδες ε, οργανωμένου εγκλήματος είναι πολύ τομεακής. Μπλέκονται σε μεγάλη ποικιλία επιχειρησιακών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτες με τεράστια προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις ευκαιρίες που αναδύονται και τις αλλαγές των περιβάλλων. Η χρήση ε, σωματικής βίας έχει αυξηθεί έντονα, ειδικότερα σε σχέση με την διακίνηση ναρκωτικών ή τα οργανωμένα εγκλήματα. Η διαφθορά είναι βασική πτυχή σε, στο οργανωμένο έγκλημα υψηλού επίπεδου. Ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος υψηλού ε, επίπεδου ε, υπησέρχονται σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς οργανισμούς χρησιμοποιώντας εκφοβισμό, απειλές και διάφορα άλλα μέσα. Οι περισσότεροι οι ύποπτοι που εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να είναι το 65% αυτών πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δομή των ομάδων οργανωμένου εγκλήματο είναι πολύ οι περισσότερε οργανώσεις είναι ε, οργανώσεις top-down, πολλά εγκλήματα γίνονται με συνεργασία στο πλαίσιο αλυσίδων συνεργασία ή οδών εμπορίας ε, με κοινή επιμελητία και με τη διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, ας δούμε την επιχείρηση Icebreaker, κοινή έρευνα διετής, στην οποία συμμετείχαν πολλέ χώρες Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία και ε, Ηνωμένο Βασίλειο με την υποστήριξη της Ευρωπόλ και της Eurojust. Το κέρδος αυτού του εγκληματικού οργανισμού εκτιμάται ότι ήταν 603 εκατομμύρια ευρώ. Τέσσερις εγκληματικές ομάδες με άνω των 50 μελών εμπλέκονταν στην διακίνηση ναρκωτικών και τσιγάρων, δολοφονίες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και λαθρεμπορία όπλων. Η έρευνα εστιάστηκε σε ένα εγκληματικό δίκτυο που υπήρχε για πολλά χρόνια με πολλά ενεργά μέλη. Η δράση έλαβε χώρα το Μάιο του 2019. 22 ύποπτοι συνελήφθησαν, 40 έρευνες πραγματοποιήθηκαν. Η αστυνομία κατάσχεσε σημαντικά χρηματικά ποσά η, εγκληματική ομάδα που καταλήθηκε είχε διακινήσει κοκαίνη από την Νότια Αμερική στη Ρωμανία. Ένα, ε, μια αποστολή, για παράδειγμα, που περιείχε 2,4 τόνους, κατασχέθηκε και οι κύριοι δράστες ε, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ξέπλυμα χρήματος. Τα μετρητά είναι ε, η σημαντικότερη απειλή στο ξέπλυμα χρήματος. Και σίγουρα αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του εγκλήματος στους υπηρεσία. Και η κατάχρηση των νέων μεθόδων πληρωμή, όπω είναι το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα γενικώ, είναι μια ανερχόμενη απειλή σε ό,τι αφορά την νομοποίηση παρανομών εσόδων. Και το τελευταίο μου σημείο αφορά την παιδική πορνογραφία και τι επιχειρήσει μα. Ε, η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο είναι σημαντική εγκληματική απειλή. Γίνονται σημαντικές σημαντικές αποσύρσεις περιεχομένου γιατί έχουμε εθνικά ε, κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2019 λάβαμε 272.000 ε, τέτοιες αιτήσει για απόσυρση περιεχομένου από το διαδίκτυο και φέτος αναμένεται να διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός των ετοιμάτων. Και μάλιστα φέτος ε, οργανώσαμε την έκτη ομάδα δράσης για τον εντοπισμό των θυμάτων με συμμετοχή 43 εμπειρογνωμόνων από 24 χώρες και 29 οργανισμούς. Και είχαμε 800 τέτοιε υποθέσεις εντοπισμού θυμάτων και εντοπίσαμε 28 θύματα και 18 αυτούργους. Σε ό,τι αφορά τι ε, μελλοντικέ απειλέ, καταρχήν σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, που είναι μια ουσιαστική απειλή στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαίου πολίτε, που επηρεάζονται όλο και περισσότερο και πλήττονται από τέτοια οργανωμένα εγκλήματα. Έχουμε αύξηση τη βία και συγκρούσει μεταξύ των εγκληματικών ομάδων. Είχαμε στη Σουηδία και Δανία τέτοιε δολοφονίε από συμμορίε και τη δολοφονία ενό. Ε, ποινικού, δικηγόρου ποινικού δικαίου στην ε, Ιρλανδία. Και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες ε, διαπιστώσαμε αύξηση της άφηξης ε, μεταναστών στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό με βάση την πείρα μας οδηγεί σε ενίσχυση του, της λαθροδιακίνησης μεταναστών και έχουμε πρωτογενείς και δευτερογενείς μετακινήσεις και συναφείς ε, απάτες. Επίσης, ε, ανησυχητική είναι η χρήση της, ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους τρομοκράτες και τις πύρες οργανωμένου εγκλήματος, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά να χρησιμοποιούν και ε, να αξιοποιούν τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτό έκαναν οι τρομοκράτε. Επίση, ε, διαπιστώνουμε αυξημένη χρήση του σκοτεινού διαδικτύου, του Darknet. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Προσπάθησα να είμαι συνοπτική στο λίγο χρόνο που είχα. Σα ευχαριστώ, κυρία Ντεμπόλ. Και όπω σα είπα, προβλέπετε συζήτηση μετά από κάθε παρουσίαση. Έχουμε εδώ ειδικά δελτία για να ζητάτε το λόγο με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το κάθε τμήμα της συνεδρίασης. Οπότε στείλτε τα στη γραμματεία παρακαλώ συμπληρωμένα αυτά τα δελτία για να ξέρουμε ποιοι θέλουν το λόγο και ποιοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε λάβει δύο γραπτές ε, προτάσεις από δύο αντιπροσωπείες πολύ πριν τη συνεδρίαση ε, για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Και με αυτές τις αντιπροσωπείες θα ξεκινήσω. Θα δώσω πρώτα το λόγο για να μας παρουσιάσει τις γραπτές, τις προτάσεις, για την της, της Γερμανικής Βουλής πρώτα και της Κυπριακής Βουλής. Θα ξεκινήσουμε με, τον εκπρόσωπο, με την εκπρόσωπο τη, του Bundestag, την κυρία Σουζάνε Μίτακ, και της δίνω κανένα δυο λεπτά για να μας παρουσιάσει αν θέλει τη γραπτή πρόταση που έκανε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή εν ώψη της συνεδρίασής μας. Είστε εδώ. Παρακαλώ κυρία Σουζάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον λόγο και ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό το οποίο μας είπε η κυρία Ντεμπόλ. Μας ανησυχεί ο προϋπολογισμός γιατί πάρα πολλά από αυτά τα οποία αποφασίσαμε και είναι απολύτως αναγκαία πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα μέσα και βλέπουμε πως ο προπολογισμός του 2020 έχει ήδη ένα έλλειμμα 30 εκατομμυρίων ευρώ και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εν μεταξύ είναι γύρω στο 50% κάτω από το απαιτούμενο ποσό και η Κομισιόν επίσης συζήτησε να μειωθούν οι θέσεις ε, στην ε, Europol οπότε το ερώτημα είναι ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Η Europol δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Όπως είπατε έχει πολλά πράγματα να κάνει και κινδυνεύει να μην ε, μπορέσει να εκτελέσει το έργο της εάν δεν υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση. Σα ευχαριστώ. Τώρα ακούσουμε... Προτείνω να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου που εκπροσωπεί την αντιπροσωπεία τη Βουλή τη Κύπρου. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη, έχετε το λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Thank you. Κύριε και κυρία Συμπροέδρη, κυρία Γενική Διευθύντρια, θα ήθελα ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας να σας ευχαριστήσουμε για τον σχολιασμό των θέσεων που έχουμε αποστείλει γραπτός. Επίσης, ε, θέλω να υπογραμμίσω τον πολύ επιτυχημένο θεσμό των guest officers. Είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη Παρασκευή να συναντηθούμε με το κλιμάκιο της Κύπρου και να δούμε η ε, διεισόμαση την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια δέχεται τις περισσότερες μεταναστευτικές ροές, δέχεται τους περισσότερους μετανάστες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο με τον μη έλεγχο των κατεχόμενων περιοχών της χώρας, και με το τι η Τουρκία στρατηγικά κάνει και το ξέρετε κύριε Αντεπόλ. Έχετε αποδείξεις από τους guest officers ότι στέλνονται οι μετανάστες με αεροπλάνα στο παράνομο αεροδρόμιο στα, στην Λευκοσία, στην, στην κατεχόμενη Λευκοσία και από εκεί διαμέσου της νεκρής ζώνης, της, της ζώνης που ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, το έδαφος της Κυπριακής, που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται άσυλο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να δούμε κατά πόσον σας ανησυχεί, κατά πόσον με την βοήθεια των guest officers που έχετε στην Κύπρο και επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν, μπορεί η Europol να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δημητρίου. Θα έλεγα τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο σε όσους το ζήτησαν. Όπως σας είπα, θα δίνω πρώτα λόγο για δύο λεπτά το πολύ πρώτα σε δύο εθνικούς βουλευτές και μετά σε έναν ευρωβουλευτή. Και μετά ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων θα ακούσουμε τις απαντήσεις από την κυρία Ντεμπόλ. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κελέτσι, από τη Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Κελέτσι, κάπως έτσι, όπως το προφέρει ο Πρόεδρος, είστε εδώ. Πέρα σας κύριε Πρόεδρε και κυρία Συμπρόεδρε. Ε, θα ε, είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπροσωπώ την περιφέρεια του Εύρου. Ο Εύρος είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Εύρος είναι μια κριτική περιοχή που συνορεύει με χερσαία και θαλάσσια σύνορα ε, με την Τουρκία. Πρόσφατα η κυρία Ντεμπόλ είχε επισκεφθεί την Άνοιξη, την περασμένη Άνοιξη, τον Εύρο και είχε διαπιστώσει ε, η ίδια το πρόβλημα των ροών που υπάρχουν, των μεγάλων ροών από τον, των μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας. Τε, τις τελευταίες μέρες πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί και οι πληθυσμοί αυτοί έχουν μεγαλώσει. Κατά την επίσκεψή της εκεί είχε τεθεί το ζήτημα της ε, τοποθέτησης guest officers και στον Εύρο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, πόσο έχει σημειωθεί, ε, κάποια, αν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ε, στο θέμα αυτό και αν προτίθεται πράγματι η Europol να τοποθετήσει guest officers στον Εύρο, καθώς επίσης να ρωτήσω για το θέμα της εξέλιξης και αν υπήρξε κάποια πρόοδος σε σχέση με τη συμφωνία της Europol και της ε, Τουρκίας ε, για την συνεργασία μεταξύ των δύο, του οργανισμού και της χώρας αυτής, ε, σε σχέση με την παροχή πληροφοριών για τα θέματα της μετανάστευσης και, του, και των εγκλημάτων με τα οποία ασχολείται η Europol. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Στρόγκσβιστ από τη Σουηδική Αντιπροσωπεία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπόλα και τους ε, εκπροσώπους της. Έχετε συνεργαστεί με τις Σουηδικές Αρμόδιες Αρχές ε, και Ε, και εκπρόσωποι του Σουηδικού Κοινοβουλίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ευρωπόλ και πιστεύω και άλλες αντιπροσωπείς θα έπρεπε να επισκέφτονται την Ευρωπόλ διότι έτσι μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τη δουλειά της Ευρωπόλ και να αναγνωρίσουν πόσο σημαντική είναι η στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των εθνικών αρχών. Αυτό το προγραμματικό έγγραφο του 2020-2022 αναφέρει το ρόλο και τις διάφορες διαδικασίες όπως αναλύσατε και εσείς. Όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν με τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Ευρωπόλια για το 2020+. Και σκέφτομαι όσον αφορά το συντονισμό και το να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες που έχουν οριστεί, είναι σημαντικό να συμφωνηθούν οι στόσεις της προτεραιότητες της στρατηγικής 2020+. Επίσης είναι σημαντικό το πώς θα μπορέσει να βρεθεί σε θέση να επιτελέσει τα καθηκοντά της Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ πιστεύω θα πρέπει να έχει συνεργασία και με την ΠΕΣΚΑ. Σε πολύ συγκεκριμένους τομείς ε, θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Την ομάδα αυτή. Ομάδα αυτή επίσης θα πρέπει λοιπόν επίσης να μας απασχολήσει το κατά πόσο μπορεί να ενισχυθεί αυτός ο συντονισμός, ούτω ώστε η Ευρωπόλ να μπορέσει να συμβάλλει πιο ενεργά. Το θέμα είναι επίσης και πώς θα αντιδράσουμε στις μελλοντικέ προκλήσεις. Για μας ε, είναι σημαντικό και από πλευρά σου ειδική αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στρόμσκβιστ. Εκπρόσωπος τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου έχει το λόγο, κύριος Αρσαλέχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την εκτελεστική διαθήκη τη Ευρωπόρ, την κυρία Ντεμπόλ, για την παρέμβασή τη και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αφοσίωσή σα στα θέματα αυτά. Όπω ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ενίσχυση και σύσφυξη των σχέσεων με την Europol και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Europol. Ε, και αυτό αντικατοπτρίστηκε ξεκάθαρα στη θέση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρηματοδότηση της Ευρωπολ στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυξάνονται τα αιτήματα προς τη Europol. Υπάρχει μια εξαιρετική αύξηση και δεν πρόκειται να μειωθεί αυτή η τάση. Και γι' αυτό, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του έργου ε, της Europol, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητε τη. Και γι' αυτό θα πρέπει να αποτρέψουμε την περικοπή στον προπολογισμό της Europol, γιατί θα έχει με τέτοια περικοπή πολύ αρνητικέ συνέπειε στο έργο αυτής τη υπηρεσία. Και είναι σημαντική και η μεικτή μας ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου για να διατρανώσει αυτό το μήνυμα και να το διαβιβάσει και στις διάφορες ε, εθνικές κυβερνήσεις για να μην γίνει περικοπή του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ. Σε περίπτωση που έχουμε το χειρότερο δημοσιονομικό σενάριο για την Ευρωπόλ, Πώ θα επηρεάσει ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο τι δραστηριότητε και τη δομή τη Ευρωπόλ και ποιοι τομεί θα επηρεαστούν κυρίω από την έλλειψη πόρων στην Ευρωπόλ. Ευχαριστούμε κύριε Σαρσαλέχο. Κυρία Ντεμπόλ. Μια και έχουμε ένα αρκετά μακροσκελή κατάλογο μελών της Επιτροπής που ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να τους ακούσουμε και να μην ξεχνούμε ότι μέχρι τις 3.30 έχουμε χρόνο για αυτό το τμήμα, για αυτή τη θεματική ενότητα της συνεδρίασής μας. Και έχουν έρθει στο μεταξύ και οι επόμενοι καλεσμένοι μας. Οπότε θα είμαστε πολύ αυστηροί πια στην τήρηση του χρόνου αγόρευσης. Και συνεχίζουμε. Θα δίνω το λόγο σε δύο εθνικού βουλευτέ και σε έναν ευρωβουλευτή και στο τέλο των ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στην εκτελεστική διευθύντρια. Η κυρία Κόνουε έχει το λόγο από την Ιρλανδία. Συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία Κόνουε, είναι ευρωβουλευτή. Πρώτα θα ακούσουμε δύο εθνικού βουλευτέ, όπω είπα. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Καλάιεν από την Ιρλανδία. Παρακαλώ. Κύριο Καλάιεν, μήπω δεν είπα σωστά το όνομά σα. Αν το κατακρεούργησα, σα ζητώ συγγνώμη και <laughs> κλιπαρώ την κατανόησή σας μικρόφωνο Mike, it's important for the translator. Είναι σημαντικό να ανάβετε το μικρόφωνο σας για να σας ακούν οι διερμηνείς και να μπορούν να σας μεταφράσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Εκτελεστική Διευθύντρια. Δεν σημείωσα στην έκθεσή σας, δεν διαπίστωσα καμία μνήμα του Brexit σε αυτά που μας είπατε και στην παρουσίαση που κάνατε. Ούτε από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο έγινε κάποια τέτοια ανοίξη από την Ευρωπόλ, αλλά δεν βλέπω και τίποτα για το Brexit στο προγραμματισμό για το 2020-2022. Λίγο πάνω από πέντε εβδομάδες μας χωρίζουν από την πιθανή άτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μπορείτε να μας ε, συμβουλεύσετε πώς ετοιμάζεται η Ευρωπόλ για τη νέα σχέση που θα έχει με το Ηνωμένο Βασίλειο όπω και να αποχωρήσει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει, για την, ε, για την αστυνομική υπηρεσία της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να συμμετέχει αμέριστα στη διομή της Ευρωπόλ και ποια θα είναι η συνεργασία ε, με την ε, αστυνομική υπηρεσία στη Βόρεια Ιρλανδία σε περίπτωση που η αστυνομία τη Βορείου Ορλανδίας ε, εξοβελιστεί από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, από την οικογένεια της Ευρωπόλ, Ποιε θα είναι οι σχέσει τη δική μα αστυνομία με την αστυνομία τη Βορείου Ορλανδίας. Τι βήματα έχουν γίνει, μπορείτε να μα ε, διαφωτίσετε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα που θα ανακύψουν εν ώψη του Brexit. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λάνετ από την Εσθονία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την ε, κυρία Ντεμπόλ για την ομιλία της και θα ήθελα να την ε, ευχαριστήσω γιατί ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστική και άρτια η παρουσίασή της. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπόλ στα θέματα της συγκέντρωσης των πληροφοριών και είπατε ότι έγινε η μετάβαση από τη συγκέντρωση δεδομένων στη συγκέντρωση πληροφοριών. Συμφωνώ μαζί σας και μετά την 20η ε, πείρα μου στην αστυνομία. Η πληροφορία έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στην διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων. Δυστυχώ γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες μέλη ακόμη δεν επενδύουν επαρκή κονδύλια στην συγκέντρωση πληροφοριών και στη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στη βάση δεδομένων της Ευρωπόλ. Αυτό βέβαια οφείλεται στα κράτη-μέλη. Αλλά αν είναι λυπή η δράση των κρατών μελών, δεν θα μπορέσει και η Ευρωπόλ να επιτελέσει το έργο της. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει και η Ευρωπόλ από πλευρά τη για να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν πιο ενεργά στη, στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων της Ευρωπόλ. Ο κύριος Βίριτανοφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Τεμπόλ για την πολύ κατατοπιστική της παρουσίαση έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Με ενδιαφέρει η συνεργασία της Ευρωπόλ με τις τρίτες χώρες. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις, ε, οι βασικές προτεραιότητες και οι δυνατότητες που έχουμε σε αυτά τα θέματα συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερω γιατί δεν εκπροσωπώ μόνο την Βουλγαρία και όχι την Εστονία, όπως είπε ο Πρόεδρος, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η γεωστρατηγική και ε, γεωπολιτική θέση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και όπως ξέρετε, η συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια ε, είχε λάβει μεγάλη σημασία όταν κορυφώθηκε ε, η τελευταία μεταναστευτική κρίση που είχαμε το 2015-2016. Και τώρα ήρθε η σειρά της κυρίας Κόνγουέι από την Ιρλανδία, του κυρίου Κόνγουέι. Κύριος είναι, είμαι, όχι κύριε. Α, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ. Ε, έλαβα μέρος σε πολλές συνεδριάσεις αυτών των επιτροπών και αυτής της ομάδας και θα θυμάστε κυρία Ντεμπόλ ότι είχα μιλήσει εκτενώς μετά το συνάδελφο Κάλλαν και εγώ για το Brexit και τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit στην Ιρλανδία, στη δική, μου, στη δική μας πατρίδα και η αυξανόμενη απειλή του Brexit και οι επιπτώσεις που θα έχει στην ασφάλεια μας ε, ανησυχούν ιδιαίτερω. Κυρία Ντεμπόλ, μα είπατε ότι θα έρθετε στο Δουβλίνο και θα μιλήσετε στην αρμόδια επιτροπή. Και μάλιστα ανταλλάξαμε και στοιχεία μετά τη συνάντηση που είχαμε στο Βουκουρέστι. Το γραφείο σας όμως, κυρία Ντεμπόλ, ούτε καν ε, ε, δεν επιβεβαίωσε την παραλαβή των mail που στείλαμε. Είναι πολύ σημαντική η μεικτή αυτή ομάδα, γιατί είναι ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω το αίτημά μου, ε, κυρία Ντεμπόλ, να έρθετε στην Ιρλανδία, να έρθετε στο Δουβλίνο και να μας μιλήσετε για αυτό το κατεπήγον ζήτημα της συνέπειας του Brexit. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κατηρός από την Κύπρο. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κυρία Ντεμπόλ, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών και ίσως νέα είδη ναρκωτικών. Στην Κύπρο είχαμε τον περασμένο μήνα μια γυναίκα νεκρή, η οποία συμμετείχε σε παγανιστικές θρησκευτικέ τελετές με χρήση ναρκωτικών, τις οποίες φέρεται να οργάνωσε αυτές τις τελετές, άνθρωπος που ήρθε στην Ευρώπη από την Κολομβία. Μετά το περιστατικό διέφυγε από την Κύπρο, νομίζω κάπου στην κεντρική Ευρώπη και είναι άφαντος. Παρακαλώ στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών διαμέσου της Europol σε ό,τι αφορά τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος θα ήθελα να μας πληροφορήσετε για τη στρατηγική σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και τον εντοπισμό διακινητών. Σας ευχαριστώ. Mrs. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τις στρατηγικές προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα εκεί που μιλήσατε ε, για το ότι ε, από πάροχος υπηρεσίας ε, στις διοκτικές αρχές θα περάσετε σε μια λειτουργία επεξεργασίας γνώσεων. Ε, θα είναι δικές σας γνώσεις ή θα είναι σύνθεση πληροφοριών από υφιστάμενες πηγές. Και μετά η στρατηγική εφισταμενες πηγες και μετα υπαριθμών 4, ότι η Europol θα είναι στην εχμή της καινοτομίας και της έρευνας. Πώς θα γίνει αυτό ε, όσον αφορά και την εμπλοκή του δημοσίου τομέα ειδικά ε, για το πώς θα διαχειριστείτε τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από ιδιωτικές εταιρείε. Και τέλος αυτό που με απασχολεί είναι η εξωτερική στρατηγική και η απόσπαση και η μετάθεση προσωπικού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ε, συνεχίζεται επί σειρά ετών. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα προσωπικού που έχει ήδη μετατεθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι αποστολές έχουν, τι ε, πληροφορίες περί απειλών συνέλεξαν και ιδιαίτερος είμαι περίεργη για τον τομέα συλλογής ε, πληροφοριών σε τρίτες χώρες. Αυτό γίνεται κατά περίπτωση ή ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνεται Σα Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιανακόπουλος τώρα από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η εμβάθυνση της συνεργασίας της Europol με τη Frontex για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στοχευμένη δράση κατά των εγκληματικών ομάδων και των τρομοκρατών είναι επιβεβλημένη. Ειδικά για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια νέα έξαρση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τα ανατολικά της σύνορα με ευθύνη της Τουρκίας. Εκατοντάδες είναι οι νεοεισερχόμενοι καθημερινά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και από την περιοχή του Εύρου στη Θράκη. Το Σάββατο στην Ελλάδα υπήρξε έκτακτη σύγκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνα υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Η κατάσταση στα νησιά είναι εκρηκτική, ενώ και στην υπηρετική Ελλάδα ασφιχτιούν τα hot spots προκαλώντα έντονε αντιδράσει στις τοπικέ κοινωνίε. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται συντονισμό Frontex και Europol για την αποκάλυψη και εξάλληψη των διεθνών κυκλωμάτων μεταφοράς και εκμετάλλευσης των μεταναστών. Ο ρόλος της Frontex δεν μπορεί να είναι η απλή καταγραφή των ισροών, ούτε είναι επιτρεπτό να αγνοείται η έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι των χωρών που έχουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή θα έπρεπε μάλιστα να διευρυνθεί και στα θέματα διακίνησης όπλων, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία. Κοινό μα στόχο δεν πρέπει να είναι άλλο από μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη συμφωνία τη Europol με την Τουρκία. Δυστυχώ, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν έχει σημειώσει πρόοδο με ευθύνη τη Τουρκία, που απαιτεί την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, στην Τουρκία δραστηριοποιείται μεγάλο αριθμό εγκληματικών οργανώσεων, κυρίω στον τομέα τη διακίνηση μεταναστών και το επίπεδο τη υφιστάμενη συνεργασία δεν επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση και εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που δρούν, εντός, ε, που δρούν εκτός, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Τουρκίας απειλεί ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη. Τι προτίθεστε λοιπόν ε, να πράξετε για την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Europol με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Onorevole Chinici del Parlamento Europeo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντεμπόλ, με την οποία έχουμε συναντηθεί επανειλημμένω εδώ. Σα ευχαριστούμε για την παρουσίασή σα και σα ευχαριστούμε που υπενθυμίσατε πόσο σημαντική είναι η JPSG για την οικονομική στήριξη τη Ευρωπόλ. γιατί αυτή η μείωση του προπολογισμού μας ανησυχεί ιδιαίτερα δεδομένων των δραστηριοτήτων που έχει να επιτελέσει η Ευρωπόλη και θα ήθελα να σας ρωτήσω επ' αυτού δύο πράγματα ε, πιο συγκεκριμένα. Εσεί, προηγουμένω, αναφερθήκατε σε αύξηση της βίας. Αναφερθήκατε επίσης και σε εγκληματικές οργανώσεις που προφανώ ε, διαχειρίζονται σημαντικά εγκλήματα, εγκλήματα για το πούμε έτσι, ναρκωτικά, οικονομικά εγκλήματα, ε, διακίνηση ανθρώπων και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν μιλάτε για οργανωμένο έγκλημα, η Ευρωπόλ διαθέτει επαρκή ε, εργαλεία και πόρους. Εσείς μιλήσατε και για νέα νομοθεσία ως προτεραιότητα. Θεωρείτε ότι χρειάζονται νέα νομοθετικά μέτρα επίσης. Επίσης όσον αφορά την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, Ξέρουμε ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να παρακολουθούνται οι χρηματικές ροές ε, λόγω της ανακύκλωσης, ε, ε, του ξεπλήματος, των κρυπτονομισμάτων, πολύ εξελιγμένων τεχνολογιών που δυσκολεύουν την ανείχνευση των χρηματικών και οικονομικών ροών. Αναφερθήκατε εσείς στο κέντρο αντιμετώπισης χρηματοοικονομικού και οικονομικού αγκλήματος Ευρωπόλ. Δεδομένων αυτών θεωρείται ότι δεδομένων και των πρόσφατων οδηγιών που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τις δραστηριότητες των αρχών επιβολής του νόμου που θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση ότι έχει αρκετά εργαλεία η Ευρωπόλ δεδομένου ότι θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία και η Ευρωπαϊκή Εισηγελία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Έμερ από την Γερμανία. Θες. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ντεμπόλ, είπατε πολύ σωστά ότι η Ευρωπόλ πρέπει να γίνει κόμβος πληροφοριών, το είπατε ρητά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αν θέλουμε τέτοιο κόμβο χρειάζονται δεδομένα και οι νόμοι προστασίας των δεδομένων στα ε, κράτη-μέλη είναι διαφορετικοί. Μελικές φορές ε, οι νόμοι έχουν τάση να ε, βοηθούν τους δράστες. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη, ποιε ε, χώρες κατά την άποψή σα μπορούν να παρέχουν τέτοια δεδομένα σωστά. Επίσης ε, αναφερθήκατε στο Brexit, ε, αναφερθήκε ο συνάδελφος από την Ιρλανδία. Αν γίνει το Brexit, ξέρουμε ότι η Αγγλία θα γίνει τρίτο κράτος μέλος τα δεδομένα που, θα, που είναι αποθηκευμένα αρχή θα μπορεί, θα να τα στείλει. Και το τρίτον, είπατε πολύ σωστά ότι είναι σημαντικό θέμα η παιδική πορνογραφία, το darknet και το ερώτημα είναι υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες να βρει κανεί ε, αυτούς που βρίσκονται από πίσω. Μπορεί η Ευρώπη μέσω υπηρεσιών Messenger, ε, μέσω διαφόρων άλλων μέσων να ε, παρακολουθεί ε, να βρει να βρίσκει ε, τους ανθρώπους που υπάρχουν, τι πρέπει να αλλάξουμε για όλα αυτά. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε να βρίσκουμε την παράνομη κατοχή ε, αγορών, αγαθών και να, αυτός που, να πρέπει αυτός που τα έχει να αποδείξει πώς τα απέκτησε. Το Ποθενέσκες δηλαδή και η Ευρωπόλ τι θα κάνει για να μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις παράνομες και να σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πόρα από την Φιλανδία. το είπα το όνομά Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας ε, εκτελεστική διευθύντρια για την ε, παρουσίασή σας. Το σχόλιο μου είναι το ίδιο με την αντιπροσωπεία που μίλησε πριν ε, φορά, τον προϋπολογισμό της Europol. Όπως όλοι ξέρουμε υπάρχουν κάποια ζητήματα πιεστικά όπως οι μεταναστευτικές ροές, τρομοκρατία, κυβερνοέγκλημα κτλ. Και ταυτόχρονα η Europol έχει αναλάβει εντελώ νέα καθήκοντα που αφορούν το λαθρεμπόριο, το κυβερνοέγκλημα και τα σχετικά. Πολλά από αυτά τα ζητήματα δεν ε, λύνονται αλλά επιδεινώνονται. Οπότε η απλή μου ερώτηση ως προς αυτό είναι αφού όλοι ε, συμφωνούμε ότι θα πρέπει η Europol να ενισχυθεί με το απαραίτητο επίπεδο πόρων. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν υπάρχει πραγματική απειλή το πολύ σημαντικό αυτό όργανο να λαμβάνει όλο και περισσότερα καθήκοντα αλλά να μην έχει επαρκείς πόρους για να τα επιτελέσει. Και αν γίνεται κάτι τέτοιο, πώς ακριβώ δίνεται προτεραιότητα σε κάποια από αυτά. Η κυρία Κένκο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Πέρσι ένας συνάδελφος από το κόμμα μου συνέταξε την, αποκάλυψε τη σχετική έκθεση για την τρομοκρατία. Μία σύσταση έλεγε πως η Europol θα πρέπει να αποτελέσει τον κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών για τα ζητήματα αυτά. Μιλάμε για πληροφορίες όπως παραδείγματος χάρη ε, λεπτομέρειες του ατόμου, βαθμός ε, ριζοσπαστικοποίησης, ε, ή εάν είχε παρελθόν με κάποια άλλα άτομα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Έχει αλλάξει κάτι έκτοτε. Έχετε ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες, υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάποια προβλήματα με την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τώρα είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, ασφάλειας και του σεβασμού των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας. Ε, δηλαδή χρειάζεται πράγματι περισσότερη προσπάθεια εδώ πέρα στην τρομοκρατία, αλλά έχουμε και άλλα εγκλήματα όπως η κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, η έλλειψη της ε, καινοτομία για να αντιμετωπίσουμε τους εγκληματίες που κρύβονται και είναι ανώνυμοι μέσω κρυπτογραφίας. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σας, να, να μου πείτε πώς είναι η δική σας η άποψη, πώς βλέπετε το μέλλον και πώς η Europol θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, εάν παραδείγματο χάρη να έχει και περικοπές στο προσωπικό. Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω πώς έχει η ισορροπία των φύλων ε, εντός της Europol όσον αφορά τις γυναίκες στα υψηλά αξιώματα. Γιατί έχει και αυτό βεβαίως την σημασία του. Σας ευχαριστώ, κυρία Μυριέντους, από, ε, από την Κύπρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχει εκτιμηθεί το ύψος των συναλλαγών που γίνονται σε κρυπτονόμισμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, κυρίως με χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Επίσης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο νομίζετε ότι χρειάζεται οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση από τα κράτη-μέλη για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ή ακόμα και της πλήρης απαγόρευσης των κρυπτονομισμάτων. Ευχαριστώ. Mr. from Belgium. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, ομάδα μας. Θεωρώ ότι η κοινή δράση Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ επικοδομητική, ειδικότερα ενώπιον ενός τόσο σημαντικού οργανισμού όπως η Ευρωπόλ. Οπότε καλωσορίζω όλους τους συναδέλφου από τα κράτη-μέλη. Έχω δύο ερωτήσεις προς την κυρία Ντεμπόλε. Πρώτον, όσον αφορά την εξωτερική στρατηγική της Ευρωπόλ και το γεγονός ότι θα συνάψει ε, συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες ή έχει ήδη συνάψει σε επιχειρησιακό επίπεδο που μερικές φορές δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, το αντικείμενο και το σκοπό και ξέρουμε ότι κάποιες από αυτές τις τρίτες χώρες μερικές φορές είναι αυταρχικά καθεστώτα. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια μέσα έχουμε για να ελέγχουμε την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών, αξιολογώντα το πώ επηρεάζουν, για παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συμφωνίε αυτέ. Και θέλω να μου πείτε και δύο λόγια παραπάνω για τι τρέχουσε διαπραγματεύσει με τι χώρε ΜΕΝΑ. Και αυτό με ενδιαφέρει. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τη συνεργασία με την Frontex. Έχει συναυθεί τον περασμένο Ιούνιο συμφωνία συνεργασία και θέλω να μου πείτε δύο λόγια παραπάνω για το αντικείμενο τη συνεργασία αυτή. Αν θέλετε μπορούμε να στείλουμε και γραπτός ε, την ερώτηση για να λάβουμε κάποιες ε, παραπάνω πληροφορίες από τη συμφωνία που βλέπουμε απλά στην ιστοσελίδα. Αν ε, αυτό είναι δυνατό πείτε μας το. Κυρία Μπρικμόντε, μόλις λάβαμε μια επιπλέον αίτηση ένα αίτημα για να πάρει κάποιο τον λόγο. Θα κλείσουμε το γύρο αγορητών με τον κύριο Ραγκούση από την Ελλάδα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, αν ακούσαμε καλά το όνομα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατά, κατά παρέκκληση, κατά κάποιο τρόπο, δυνατότητα να, πω δύο, να θέσω δύο θέματα. Το ένα κυρίως για να ε, ενισχύσουμε και εμείς ε, την, ε, τον πολύ σοβαρό προβληματισμό που ε, βάσιμα αναπτύχθηκε σχετικά με τον προϋπολογισμό που θα στηρίξει οικονομικά τις δραστηριότητες της Europol. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι σήμερα, δεδομένου ότι έτσι και αλλιώς για τα θέματα του προσφυγικού και της όξυνσης που έχουμε στις ροές αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι και από το Ελληνικό και από το Κυπριακό Κοινοβούλιο, σήμερα ε, διεξάγεται στον ΟΗΕ ε, η Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα. Και είναι μία από τις ε, βασικές αρμοδιότητες της Europol η δίωξη του εγκλήματος σε σχέση με το περιβάλλον. Ε, θα ήθελα αν έχει υποθεί κάτι να επαναληφθεί, αν δεν έχει υποθεί ε, τότε να λεχθεί τώρα, δηλαδή τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η στρατηγική για την καταπολέμηση του, του εγκλήματος σχετικά με το περιβάλλον, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ε, αποτέλεσμα ε, και εγκληματικών μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε, ε, πολλές, ε, σε πολλά σημεία γεωγραφικά μήκη και πλάτη και της Ευρωπαϊκής Υπήρου και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ. we've had... Ωραία. Ακούσαμε πάνω από 20 ε, ερωτήσεις. Όλες σεβάστηκαν τον χρόνο, κατά το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερος και σας ευχαριστώ. Και έχουμε γύρω στα 50, 15 ε, λεπτά Λοιπόν, ε, τα μαθαίνετε Σιγά σιγά, ε, κυρία Ντεμπόλ, σας παρακαλώ προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ για τον προπολογισμό. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες και ε, να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Λοιπόν, οι πρώτε ερωτήσει ε, για τον ε, προϋπολογισμό. Πράγματι, η πρόταση του προϋπολογισμού για το 2020 που δημοσίευσε η Κομισιόν τον Μάιο ήταν κάτω από τις προσδοκίε, Ήταν μείον 33 εκατομμύρια και μείον 50 ε, θέσεις προσωπικού ε, σε σχέση με αυτό το οποία είχε προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντα βέβαια εκτιμούμε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανησυχία μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες μαζί με τα κράτη-μέλη για να ε, γίνει καλύτερη η εξωτερική ασφάλεια. Ε, μας απασχολεί η απειλή της εσωτερικής ασφάλειας ε, και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής απειλής ασφαλείας, έτσι ώστε σε, στο επίπεδο της εσωτερικής ασφαλείας να μην είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν και αυτό το οποίο τι πρέπει να κάνουμε εάν ε, ο τελικός ε, προϋπολογισμός ε, δεν θα είναι αυτό το οποίο είχε προτείνει το ΔΣ της Europol. Θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες όπως περιγράφονται στο προγραμματικό έγγραφο και κάποιες μακροπρόθεσμες αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη στρατηγική για το 2020 και μετά. Αυτό το οποίο θα επηρεαστεί είναι η ανάπτυξη guest officers στα hotspot της μετανάστευσης. Θα επηρεαστεί επίσης η καταπολέμηση των δευτερογενών μετακινήσεων. Θα θέλαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, γιατί βλέπουμε μια αύξηση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν, αύξηση της βίας η απάντηση από την ευρωπαϊκή διάσταση θα επηρεαστεί γιατί θα πρέπει να επανεστιάσουμε τις ε, προσπάθειες σε στόχους υψηλής αξίας. Αυτό σημαίνει ότι ήδη σήμερα τώρα δίνουμε προτεραιότητα σε, ποιε, σε ποιες περιπτώσεις ε, στηρίζουμε και σε ποιες περιπτώσεις ε, δεν στηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Έχουμε λεφτά για 15 υποθέσεις μόνο για στόχους υψηλής αξίας και ε, χρειαζόμαστε 45-50 υποθέσεις να στηρίξουμε με διεπιστημονικές ομάδες ε, σε επιχειρησιακές ε, ομάδες της Europol για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Europol. Ήδη ε, δραστηριοποιούμαστε όσον αφορά τα έργα EMPAC. Έχουμε και ένα αναλυτικό σχέδιο καταπολέμησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ε, εμείς εξαρτώμαθα από την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη, αλλά και εκεί βεβαίως ε, θα επηρεαστούμε στην ε, στήριξη που μπορούμε να δώσουμε. Η επένδυση στον τομέα της πληροφορικής και το παράδειγμα του παράνομου περιεχομένου στο διαδικτύο. Πρέπει να αναβαθμίσουμε το σύστημά μας, ονόματι Ήρμα, να πάμε σε ένα πιο ευπροσάρμοστο σύστημα το οποίο θα μπορεί να αναπτυχθεί στα διάφορα κράτη-μέλη, στις μονάδες διαδικτύου. Ε, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Αν δεν έχουμε τα λεφτά από το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το σύστημα και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επενδύσει μετά μόνο του. Κάτι το οποίο ε, θα είναι κόστος για τα κράτη-μέλη αλλά και θα δυσκολέψει την ε, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως για να δίνονται οι πληροφορίες στους παρόχους. Λοιπόν, και η δική σας στήριξη είναι άρα πάρα πολύ σημαντική και για την καινοτομία και για την έρευνα. Γιατί έχουμε αυτές τις, ε, αυτή την στρατηγική προτεραιότητα για να είμαστε στην αιχμή της έρευνας. Γιατί αυτή είναι η απέτηση των κρατών μελών. Όλοι ε, έχουν την πίεση για να μειώσουν τους πόρους. Οπότε τα κράτη-μέλη, οι ιδιοκτικές αρχές προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμε λύσεις για την αστυνόμευση και τα ζητήματα ασφαλεία. Ε, από κοινού. Έχουμε τώρα ένα έργο το οποίο εξετάζει τα διάφορα βήματα που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Αξιολογούμε το τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω, γι' αυτό ε, χρειαζόμαστε προπολογισμό. Και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές αστυνομικές λύσεις για όλα τα κράτη-μέλη, για όσα έχουν τα κονδύλια και για όσα δεν τα έχουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το θέμα των αποσπασμένων αξιωματικών στην Κύπρο. Κοιτάξτε, η εντολή μας είναι σαφής, δεν είμαστε ευρωπαϊκό FBI και δεν μπορούμε να λάβουμε εκτελεστικά μέτρα. Πάντα επανερχόμαστε στην εντολή μας. Η εντολή της Europol είναι να συνδέει, να είναι ο κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών για ζητήματα σοβαρών εγκλημάτων και να σέβεται τα όσα αναφέρονται στο παράδειγμα 1 και 2 του κανονισμού μας για σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Δεχόμαστε λοιπόν πληροφορίες μόνο από τα κράτη-μέλη, μόνο όταν είναι συμβατό με το νομικό μας πλαίσιο και μετά επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ε, πάντα σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη. Πάντα λοιπόν το κράτος μέλος ορίζει το τι μπορεί να κάνει η Europol με τις πληροφορίες που μας δίνει. Δηλαδή, αν μας πει ότι αυτό το στέλνουμε μόνο για διασταύρωση, το, το χρησιμοποιούμε μόνο για διασταύρωση αν μας πει μπορείτε να το επεξεργαστείτε και ε, να δώσετε νέα πηγές στους ερευνητέ. Αυτό κάνουμε. Οι πληροφορίες ε, παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών. Η Europol δεν είναι ο ιδιοκτήτης ε, των πληροφοριών αυτών τα κριτήρια τώρα στην περίπτωση της ε, Κύπρου. Είχαμε ένα ζήτημα γιατί ακριβώς ε, επειδή δίνουμε κάποιες προτεραιότητες δεν ε, μπορούμε να στηρίξουμε επαρκώς τις κυπριακές αρχές γιατί έχουμε το κριτήριο με βάση τον πληθυσμό. Αλλάξαμε τα κριτήρια, γνωρίζαμε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές διοκτικές αρχές και τώρα έχουμε την δυνατότητα να στηρίξουμε τις κυπριακές αρχές καλύτερα και περισσότερο από ό,τι πριν αλλά εξαρτάται από τις κυπριακές αρχές ε, το να φέρουν υποθέσεις και μετά μαζί με τον ε, σύνδεσμο στη Χάγη να αξιολογήσουμε την ε, δυνατότητα στήριξης των κυπριακών αρχών στις διάφορες υποθέσεις. Εστιάζουμε στη διακίνηση ανθρώπων και αυτό είναι μέρος της εντολής μας και στις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Ο συντονισμός και η συνεννόηση ε, αξιολογείται ως πάρα πολύ καλή. Ε, ο Εύρος τώρα, πράγματι επισκέφθηκα την περιοχή. Δεν στέλνουμε εκεί πέρα αποσπασμένου εξωματικού. στέλνουμε όμως αναλυτές που βοηθούν τις διοκτικέ αρχές στην επεξεργασία των δεδομένων στις ε, ποινικέ υποθέσει. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Europol, έχουμε μια στρατηγική συμφωνία με την Τουρκία. Υπάρχει ένα σύνδεσμος από την Τουρκία στο αρχηγείο, στην Europol, αλλά δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να ανταλλάξουμε επιχειρησιακά δεδομένα με την Τουρκία, γιατί δεν έχουμε επιχειρησιακή συμφωνία. Η Κομισιόν λοιπόν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή μια επιχειρησιακή συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει εδώ πέρα ένας ρόλος ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις τέτοιων συμφωνιών, ε, κάτι το οποίο, όπως είπα, λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Η εξωτερική στρατηγική τώρα και η συνεργασία με τις ε, τρίτες χώρες, η εξωτερική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δούμε παραδείγματος χάρη το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, 65% των ε, ηγετών τέτοιων ε, εγκληματικών ομάδων ε, είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει πως οι υπόλοιποι δεν είναι. Ε, τώρα δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα πληροφοριών εάν δεν έχουμε πληροφορίες από τρίτες χώρες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε επιχειρησιακέ συμφωνίε. Όταν μιλάμε για ναρκωτικά, παραδείγματο χάρη, να έχουμε επιχειρησιακή συμφωνία με την Κολομβία και στρατηγική και επιχειρησιακή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μοιραστούμε δεδομένα με τις Κολομβιανές αρχές και να συνεργαστούμε με τουλάχιστον δύο μέλη και η Europol με την Κολομβία. Τώρα για τρίτες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε επιχειρησιακή συμφωνίες με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά πρέπει να δούμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είναι ακόμα στο κατάλληλο επίπεδο. Για εμάς είναι κάτι το σημαντικό και πολύ σημαντική περιοχή του κόσμου ε, για να έχουμε συνεργασία. Brexit. Ε, συζητήσαμε όλα τα σενάρια που αφορούν το Brexit ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζητήσαμε κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάσαμε τα διαφορετικά σενάρια και τα βήματα που θα λάβει η Europol σε σχέση με το Brexit και έχουμε διαφορετικά σενάρια για τις διαφορετικές ε, πιθανότητες, ε, για τις διαφορετικές ε, αποφάσεις που ίσως ληφθούν. Ζητώ συγγνώμη για το ότι δεν απάντησα στην πρόσκληση για να πάω στην ε, Ιρλανδία να μιλήσω στην Βουλή θα το ε, δούμε οπωσδήποτε αλλά μπορείτε πάντα να έρθετε και σε επαφή εδώ πέρα με το γραφείο μας στις Βρυξέλλες πρέπει να είμαστε και σε στενή επαφή με την Task Force 50 που αφορά ακριβώς τη συζήτηση του Brexit. Συλλογή πληροφοριών στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίσης ε, πάρα πολύ σημαντικό. Έκανα πέρσι την προσπάθεια να πάω σε όλα τα κρατομέλη, στα και να θέσω τα ζητήματα αυτά με όλους τους εταίρους για να υπάρξει αυτή η αντάλυση εις βάθος για την ανταλλαγή πληροφοριών. Γνωρίζουμε και στο μέλλον θα εστιάσουμε στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, όπως ξέρετε και για τρομοκρατία και ε, λαθροδιακίνηση μεταναστών κτλ. Πρέπει να συνεργαστούμε, να φτιάξουμε ομάδες εργασίας, να έρθουν σε επαφή οι ερευνητές και να έχουν και τις κατάλληλες πληροφορίες. Και μετά από κοινού αναπτύσσουμε ένα σχέδιο δράσης για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, διαφορετικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος η πλατφόρμα για τις ευρωπαϊκές αστυνομικές λύσεις, ε, την έρευνα και ανάπτυξη. Επειδή ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά και οι πόροι περιορισμένοι, προσπαθούμε ακριβώς ε, να συνεργαστούμε και όπου μπορούμε και η Europol είναι μια πλατφόρμα όπου οι αστυνομικές υπηρεσίες ε, να μπορούν να έρθουν σε επαφή, όπου θα έχουν μια εικόνα των εξελίξεων στις διαφορετικές χώρες για να έρθουν σε επαφή με τις χώρες αυτές για να μπορέσουν να δουν πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι τις απειλές ασφαλείας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να προσφέρουμε καινοτόμε λύσεις για τις διοκτικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Η συνεργασία με τη Frontex και τη Europol είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Πέρσι είχαμε κοινό διοικητικό συμβούλιο όπου παρουσιάσαμε ακριβώς ε, το προς τα που θα κινηθεί η μελλοντική μας συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς εν εξελίξη, η συνεργασία Frontex Europol, αλλά η εκτελεστική διευθύντρια της Frontex και εγώ βεβαίως ε, θα συνεργαστούμε και προσπαθούμε να μην κάνουμε δύο φορές τα ίδια πράγματα. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους σχετικούς κανόνες. Υπάρχουν πράγματι διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να συνεργαστούμε με το νομικό πλαίσιο που έχουμε. Και έχουμε έναν ε, αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα με 10 άτομα που κάθε μέρα αξιολογούν το πώς εργαζόμαστε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο για να εξυπηρετήσουμε τα κρατημέλη ακόμα καλύτερα. Αλλά εάν ε, ε, να γίνει μια συζήτηση εις βάθος για την προστασία των δεδομένων, ε, ευχαρίστως να λάβουμε κι εμείς μέρος και βεβαίως και το νέο νομικό πλαίσιο της Eurojust είναι πιο προσαρμοσμένο στο νέο τοπίο ασφαλείας, ε, θα έλεγα, ε, που αντιμετωπίζει και η Europol. Οι προτεραιότητες τώρα της Europol είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά. Ε, κοιτώντας ε, το οργανωμένο έγκλημα, είναι εγκληματικό δρά παγκοσμίω. Υπάρχει πλέον το έγκλημα ως υπηρεσία βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των εισαγωγών ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κόμβοι για τα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία εξάγονται σε άλλες χώρες. Πολλές από τις εγκληματικέ δραστηριότητες των ομάδων γίνονται πιο περίπλοκες και απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική και βλέπουμε την ανάγκη τη ζήτηση από τα κράτη-μέλη να περάσουμε περισσότερο στο οικονομικό έγκλημα. Γι' αυτό ακριβώς φτιάχνουμε το κέντρο οικονομικού εγκλήματος, γιατί πρέπει να είναι κανείς ειδικό σε αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να παρακολουθήσει το χρήμα και δεν έχουμε όλη την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη αυτή τη στιγμή ε, στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πρέπει να ενισχυθούμε εδώ. Οι αριθμοί δείχνουν ότι μόλις 2,1% των ε, προϊόντων εγκλήματος ε, δεσμεύονται και ένα εκατό κατάσχεται. Είναι πολύ χαμηλά αυτά τα νούμερα και πραγματικά αποσταθεροποιούν την οικονομία. Λοιπόν, ε, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου τις στείλετε εμένα και θα σας δώσουμε τις απαντήσεις γραπτός και να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε και την Europol για να συζητήσουμε εις βάθος. Σας ευχαριστούμε αγαπητή κυρία Ντεμπόλ. Κάνατε, είμαι βέβαιο ότι καλύτερο. Δεν μα εκπλήσει γιατί ακριβώ αυτό ήταν ο σκοπό μα εδώ. Έλεγχο τη Ευρωπόλη, δηλαδή ημών. Με διάφορου τρόπου. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο βήμα. Ευχαριστούμε που κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε για να απαντήσετε στι διάφορε ερωτήσει των μελών αυτές τις συνεδρίαση και τώρα προτείνω χωρί καμία καθυστέρηση, διότι έχουμε ήδη 5 λεπτά καθυστέρηση. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης χωρίς διακοπή. Στις 4 και 4 θα σταματήσουμε για καφέ μεν, απομένουν 45 λεπτά για να ακούσουμε τους επόμενους προσκεκλημένους μας, ε, τον κύριο Αντρέι Λίντα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ, την κυρία Οάννα Φλωρέα, πρώην συμπρόεδρος της ε, JPSG, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ρωμανικού Κοινοβουλίου στην JPSG, ως ε, παρατηρητής αυτή τη στιγμή συμμετέχει αυτής της μεικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου. yeah, yeah. The, the, the, I was just uh, trying to frame the, the following point by reminding you. Θα σας παρουσιάσω το επόμενο σημείο ε, λέγοντας ότι αυτό το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να υιοθετεί τον πολιετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ και τον πολιετή προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Ε, δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού της Ευρωπόλ το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε άτομο μπορεί να δώσει μια σημαντική ε, γνωμοδότηση ε, για οποιαδήποτε συζήτηση. Γι' αυτό εδώ έχουμε καλέσει τον κύριο Λίντσα και την κυρία Φλόρεα. Στην τελευταία συνεδρίαση του JPSG τον Φεβρουάριο δεν ελήφθη καμία απόφαση για το ζήτημα του εκπροσώπου του JPSG που θα μπορούσε να, παρα... να παρίσταται σε συνεδριάσεις ως παρατηρητής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ. Έτσι λοιπόν οι συμπρόεδροι εκπροσωπούσαν την JPSG και η πρώην συμπρόεδρος κυρία Φλόρεα παρέστη στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μάιο φέτος. Η κυρία Φλόρεα υπέβαλε την γραπτή της έκθεση στην JPSG πριν τη συνεδρίαση αυτή και θα μας την παρουσιάσει σήμερα εδώ αυτοπροσώπως σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και έχετε το λόγο. Έχετε υπόψη ότι συνολικά έχουμε μόνο 45 λεπτά. Και αναμένουμε ότι θα ε, γίνει και μια συζήτηση με τα μέλη πριν σταματήσουμε για καφέ. Έχετε το λόγο κυρία Φλόρεα, ο κύριος Λίντσα πρώτα και θα έλεγα 10 λεπτά καθής και το πολύ και μετά να ανοίξουμε, να δώσουμε το λόγο στα μέλη, δύο λεπτά το πολύ για κάθε ερώτηση που θα απευθύνεται στα μέλη του πάνελ. Έχετε το λόγο κύριε Λίντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της JPSG και αξιότιμα, συμπρόεδρε η κύριε Λόπες και κυρία ε, Ταλβίτη. Όπως ζητήσατε θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Θα σας παρακαλουσιάσω τις βασικές λειτουργίες του Διοικητικού Συμβούλου και τις κύριες δραστηριότητες μετά από την τελευταία συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2019. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Θα είμαι πολύ σύντομος όπως προτείνατε και θα συζητήσουμε το σημερινό και τον αυριανό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί σα, χωρί καθυστέρηση να σα πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό κυβερνητικό όργανο του οργανισμού. Εκπροσωπεί τι αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών, που είναι οι κύριοι ενδιαφερομένοι στην Ευρωπόλ. Όπω είπατε πολύ σωστά και στην αρχή, και αυτό ήθελα να ξανατονίσω, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο διακυβέρνηση τη Ευρωπόλ αποτελείται από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Την 1η Οκτωβρίου του 1998 έγινε η πρώτη συνάντηση και έκτοτε εξελίχθηκε σημαντικά το νομικό πλαίσιο της Ευρωπόλ. Σε όλο αυτό το διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο καθοδηγεί και επιβλέπει τον Ευρωπόλ σήμερα. Οι λειτουργίες στρατηγικού σχεδιασμού, ε, προγραμματισμού, ε, ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπόλ. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο υιοθετεί την πολιτική προγραμματισμό, για τον οποίο έχουμε ακούσει πολλά, το ετήσιο πρόγραμμα εργασία και τον προπολογισμό της Ευρωπόλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση τη Ευρωπόλ αλλά και τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες διορισμού του προσωπικού της Ευρωπόλ και του εκτελεστικού διευθυντή. Επίσης, καθορίζει τον αξιωματικό προστασίας δεδομένων, τον αξιωματικό ε, λογιστικής και καθορίζει και τις δυνατότητες του εσωτερικού ελεγχού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μαζί με τη γραμματεία αποτελούν τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τις επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή και υιοθετεί την ετήσια ενοποιημένη έκθεση ε, δραστηριοτήτων του Ευρωπόλ. Επίση, το Συμβούλιο ασκεί ε, ρυθμιστική λειτουργία που αφορά όλες τις δραστηριότητες και την καλή λειτουργία της Ευρωπόλ και την εκτέλεση της ε, εντολής. Για παράδειγμα, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε ε, τα δικαιώματα και τις υποχρώσεις των αξιωματικών συνδέσμων που αποσπά το προσωπικό τους κανονισμούς, τους κανόνες ε, διορισμού ε, των διευθυντών και των εκτελεστικών διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών ε, κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων των μελών και κατευθυντήρες γραμμές για την υλοποίηση των νέων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που είναι γνωστό ως σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης δεδομένων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει ότι οι πράξεις προς εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών αντιστοιχούν ε, στους σκοπούς ε, της Ευρωπόλη. απόφαση του 2016 αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 1049 κάτω 2001 του κανονισμού για τη διαφάνεια και καθορίζει τα όρια της δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα της Ευρωπόλ επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ προστασίας δεδομένων, απορρίτου, αφενός και λογοδοσίας και διαφάνειας αφετέρου. Θα αναρωτιέστε πώς λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προ... Η Πρόεδρος συγκαλεί τις συναντήσεις του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Στις 4 Οκτωβρίου εγώ θα προεδρεύσω την 112η συνεδρίαση του Συμβουλίου. Παρότι ο κανονισμό μα απαιτεί, από εμά να έχουμε τουλάχιστον δύο τακτικέ συναντήσει ετησίω, που στην πραγματικότητα συναντιέται τέσσερι φορέ ετησίω το Συμβούλιο. Αυτό πιστεύω δείχνει πόσο μεγάλο είναι ο φόρτο εργασία του. Επιπλέον, δύο ομάδε εργασία, μία για θέματα συνεργασία και το άλλο για ε, διαχείριση πληροφοριών, συναντώνται συχνά. Στην άσκηση της λήψης αποφάσεων, το Συμβούλιο βασίζεται επίση και στην συμβουλευτική υποστήριξη των άλλων φορά τη Ευρωπόλ ε, με εκπροσώπους των κρατών μελών, όπως η επικεφαλής των εθνικών ε, τμήματων ε, της Ευρωπόλ, που είναι αυτοί που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της Ευρωπόλ ή η Επιτροπή Ασφάλειας που είναι υπεύθυνη για τα πρότυπα και την τήρηση των προτύπων ασφαλείας της Ευρωπόλ τα ποικίλα θέματα με τα οποία ασχολείται το Διοικητικό Συμβούλιο αντικατοπτρίζονται και στι ημερήσεις διατάξεις των συνεδριάσεών του. Η βασική του ε, φορείς είναι τα μέλη του. Το αποτελείται από ένα μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε κράτος μέλος και από την Κομισιόν. Ιστορικά έχουμε παρατηρήσει και η εμπειρία μα μας λέει σήμερα ότι ε, οι ικανότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αφοσίωσή του είναι σημαντικοί παράγοντε ώστε η Ευρωπόλη να είναι υποδειγματικό οργανισμό επιβολή του νόμου στην Ευρώπη και παγκοσμίω επίση. Επιπλέον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων εθνικών αρχών σε επιχειρησιακό και σε πολιτικό επίπεδο μέσω επιστολών προς τα Υπουργεία Εσωτερικών. Η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση εξηγεί και το πώς λαμβάνουμε αποφάσεις. Με περηφάνεια μπορώ να πω ότι λόγω της, προσέγγισης, της συνενετικής προσέγγισης που έχουμε λαμβάνουμε αποφάσεις στο Συμβούλιο μόνο ομόφωνα. Δεν εκπλήττει λοιπόν που ουδέποτε έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο παρά τις διαφορετικές ε, ε, νοοτροπίες λειτουργούμε ως ένα συνεργατικό σώμα ενωμένο διότι έχουμε ως κύριο σκοπό να ενισχύουμε το έργο της Ευρωπόλ στις έρευνες για το διασυνορικό έγκλημα και την, και την τρομοκρατία. Φυσικά τέτοια αποτελέσματα θα ήταν αδύνατα χωρίς την προπαρασκευαστική εργασία των της Ευρωπόλ υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διευθύντριας. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου παρακαλώ να πω δύο λόγια για το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα λειτουργεί με μια περίπλοκη δομή διακυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άμεσα το έργο μαζί με την JPSG και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Ανάλογα ο καθένα με τι αρμοδιότητέ του. Ω αποτέλεσμα, από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού τη Ευρωπόλ, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ω προτεραιότητα τη διακυβέρνηση και του ελέγχου. Επιπλέον, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παίζουν σημαντικό ρόλο ως δημοσιονομικές αρχές της Ευρωπόλ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξαρτάται σε αυτό το επίπεδο από τις δικές τους αποφάσεις. Λόγω όμως της ιδιαίτερης σύνθεσης και εντολής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί ένα μοναδικό φορέα για την Ευρωπόλ. Αξιολογεί πώς επιδρούν οι νέες ε, εντολές, ε, τις δυνατότητες του οργανισμού μας, τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να σχεδιάσουμε τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες και να εκπληρώσουμε τις βασικές μας ε, εντολές προς όφελος των κρατών μελών. Εγώ από εμπειρία μου θα σας πω ότι η διαχείριση σε ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά έργα σε πρώιμο στάδιο βοηθά και τα κράτη-μέλη να είναι πιο εύκολη η υλοποίηση και η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές. Το έργο διαλειτουργικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άριστο παράδειγμα, επειδή το Συμβούλιο διαρκώ παρακολουθεί το πώ επιδρά αυτό το έργο στην Ευρωπόλ και στα κράτη-μέλη. Μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων της Ευρωπόλ, η JPSG που συνδέει τα κράτη-μέλη με την Ευρωπόλ είναι βασικός εταίρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεργασία έχει εξελιχθεί περισσότερα μετά από τη συνεδρίαση της JPSG το Φεβρουάριο δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού της Ευρωπόλ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Κάλεσα εκπροσώπους της JPSG στην τελευταία μας ε, συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι το Μάιο ως παρατηρητές. Και είχαμε τη συμπρόεδρο την κυρία Φλόρεα, η οποία συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για σημαντικά θέματα της ημερησίας διάταξης εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω την κυρία Φλόρεα για τη σημαντική τη συμβολή στι συζητήσεις μα. Η έκβαση τη τελευταία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Μάιο δείχνει πόσο πολλέ και ποικίλε είναι οι λειτουργίε του Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, υιοθετήσαμε την ετήσια ενοποιημένη έκθεση δραστηριοτήτων για το 2018 που διαβάστηκε στην JPSG και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις λειτουργίε που θεσπίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για τη ε, δημιουργία των εσωτερικών δομών τη Ευρωπόλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει λοιπόν την οργάνωση προσαρμογών δυνάμει της νέας στρατηγικής της Ευρωπόλ 2020 συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένου του νέου ε, κέντρου αντιμετώπισης χρηματοοικονομικού και οικονομικού εγκλήματο. Επίση, λαμβάνει αποφάσει σε σχέση με το προσωπικό. Όσον αφορά μελλοντικέ αποφάσει για το θέμα, το Συμβούλιο επίση συζήτησε σημαντικά δημοσιονομικά θέματα, πώ επιδρούν οι δραστηριότητε προτεραιότητα τα πράγματα και οι δυσίωνε προοπτικές για τον προπολογισμό το 2020 και η πολιετη δημοσιονομική προοπτική 2021-2027 και η επερχόμενη συνάντηση που θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα στην Χάγη και εκεί η Ευρωπόλ θα εξετάσει αυτό το ζωτικό ζήτημα από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Πριν κλείσουμε για τι τελευταίε δραστηριότητε του Συμβουλίου, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμό Ευρωπόλ, όλε οι συνόψει ε, των ε, πρακτικών των συνεδριάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπόλ. Αυτή η πρακτική συνάδει με την αρχή της διαφάνειας που ανέφερα προηγουμένως, αλλά με την επιφύλαξη ε, συνεδριάσεων ε, που μπορεί να αποφασίσουν να εφαρμόσουν το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα σε ορισμένα έγγραφα για επιχειρησιακά ζητήματα. Θα κλείσω με κάποιες παρατηρήσεις για το μέλλον. Το πολιτές πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπόλ που υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου φέτος μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θα διαμορφώσουν το έργο μας για την επόμενη τριετία δηλαδή από τα έτη 2020 μέχρι το 2022. Στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, όπως σας είπε και η εκτελεστική διευθύντρια, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτών των γράφων προγραμματισμού είναι σημαντικό και Σίγουρα τέτοιο προγραμματισμός ε, σκοπό έχει να υλοποιήσει του στόχου και τι προσδοκίε των κρατών μελών και να επιφέρει κάποια προστιθέμενη αξία στο έργο, το καθημερινό έργο των εθνικών διεκτικών αρχών, ιδιαίτερα στα θέματα διασυνοριακού εγκλήματος και τρομοκρατία. Και μάλιστα έχουμε τι στρατηγικέ προτεραιότητε με βάση τον προγραμματισμό τη Ευρωπόλ και τι δραστηριότητε που έχουν προγραμματιστεί και που είναι απολύτω απαραίτητε. Όπω φαίνεται και από τα στατιστικά αποτελέσματα που υιοθετεί η Ευρωπόλ στην έκθεση υπεπραγμένων, τα κράτη-μέλη ε, εξαρτάται όλο και περισσότερο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ευρωπόλ. Και σίγουρα η τάση αυτή θα αυξηθεί στο μέλλον, γιατί οι ιδιοκτικές και οι αρχές επιβολής του νόμου θα χρειαστούν την αφοσιωμένη υποστήριξη της Ευρωπόλ για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, όπως την ε, αύξηση νέων τεχνολογιών, όπως τις 5G, που απαιτεί περισσότερες ικανότητες και Επίση, ε, τα, μεγάλα, τα μαζικά δεδομένα δημιουργούν προβλήματα ασφάλεια και για του Ευρωπαίου πολίτε. Και αύριο ο Άνση Κάγκα από τη Φιλανδία θα σα παρουσιάσει ε, ε, τα θέματα της, του Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Συμβουλίου και πώ σκοπεύει η Ευρωπόλ να διευκολύνει το έργο των εθνικών αρχών για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα τη Ευρωπόλ. Επιπλέον, είναι σημαντικό για την Ευρωπόλα να αυξήσει τη συνεργασία και τη συνέργεια με, τις άλλες, με τους άλλους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών. Και έτσι θα, υλοποιήσουμε, θα από κοινού τους πολίτες μας στόχους και θα συσφίξουμε τους, τους δεσμούς και με τους άλλους οργανισμούς ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών και με το νέο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε ε, να έχουμε μια πολυεπίπεδη συνεργασία με όλους αυτούς τους οργανισμούς που εμπίπτουν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Αυτά ευχαριστώ και περιμένω τις απορίες σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίντσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Οάννα Κονσουέλα Φλωρέα που θα μας ενημερώσει για τη συμμετοχή της στην 110 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλης. Σας ευχαριστώ τα πολύ 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Δεν πρόκειται να διαβάσω την έκθεσή μου, γιατί την, σα την έχω διαβιβάσει. Θα κάνω μια λίγα σύντομα σχόλια. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προ τον κύριο Αντρέη Λίντσα, που με προσκάλεσε ω συμπρόεδρο τη μεικτή ομάδα για να λάβω μέρο στην 110η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπόλ. Επίση, θα ήθελα επευκαιρία να εξάρω την παγιωμένη σχέση που έχουμε αναπτύξει από την έναρξη των ανδραστηριοτήτων το 2017 ε, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Θα ήθελα αυτή εξ αρχής να επισημάνω ότι φέτος ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ ε, αύξησε τον αριθμό των σημείων ημερής της διάταξης, το οποίο μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος της μεικτής μας ομάδας. Αυτό δείχνει εμπράκτο στην εμπιστοσύνη και την ε, επικοδομητική συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι δύο φορείς μας τους τελευταίους μήνες. Βασικός μου στόχος ως εκπρόσωπος της μεικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ ήταν να δημιουργήσω στενούς δεσμούς μεταξύ του οργανισμού και της δικής μας μεικτής ομάδας και να ενημερώνω όχι μόνο για τα βασικά θέματα, αλλά και για άλλες ανησυχίες και παρατηρήσεις ε, που συζητήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση του Μαΐου, για τον προπολογισμό για παράδειγμα. Στη δική μου έκθεση που σας επέστειλα τον Ιούλιο, θα βρείτε και μία σύνοψη πολύ καρποφόρων συζητήσεων που είχα με την εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ, με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι βέβαια ότι πολλά από τα θέματα αυτά θα συζητηθούν και σήμερα, γιατί είναι κεφαλαιόδου σημασία για τη μελλοντική εξέλιξη του οργανισμού. Στι απαιτήσει και τι μεγάλε προκλήσει που δημιουργεί το κλίμα ασφάλεια στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ανοιχτού διάβλου καθ' όλη τη διάρκεια του έτου και όχι μόνο κατά τι εξάμεινε μα συναντήσει. Οπότε θα ήθελα επ' ευκαιρία να ε, χαιρετήσω τη δεκτικότητα και προθυμία των εκπροσώπων της Ευρωπόλ και ιδιαίτερα της εκτελεστικής διευθύντρια κυρίας Κατρίν Ντεμπόλ που έσπεψαν να απαντήσουν σε όλα τα αιτήματα και τις απορίες μας. Σε όλε τι παρεμβάσει μου επισήμανα ότι είναι πολύ σημαντικό για τη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου να λαμβάνει εγκαίρω όλε τι απαραίτητε πληροφορίε για να μπορέσει να ασκήσει απρόσκοπτα το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίση, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα βασικά μέσα που έχει η μεικτή ομάδα κατά την άσκηση των λειτουργιών τη ε, ε, προφορικές και γραπτές ερωτήσεις και τις ε, δυνατότητες να κάνουμε καλύτερη χρήση αυτών των μέσων. Η κυρία Κατρίντα Βόλα παρουσίασε στην ομιλία της τις βασικές προτάσεις για τις οργανωτικές αλλαγές με βάση τη στρατηγική 2020 και επέκεινα. Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Αστυνομικής Υπηρεσία. Για να προσαρμοστεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον, η Ευρωπόλ θα συγκεντρώσει όλε τι υπάρχουσε εσωτερικέ ε, δημοσιονομικέ λειτουργίε σε μια ενιαία δημοσιονομική μονάδα που θα δημιουργηθεί και θα υπάγεται στο, στη Διεύθυνση Ικανοτήτων. Επίσης, ε, σκοπεύει να και θα προσπαθήσει να απαντήσει άμεσα στα αιτήματα των κρατών μελών σε θέματα χρηματοοικονομικού και οικονομικού εγκλήματο και θα συστήσει τον Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματο που θα υπάγεται στη διεύθυνση επιχειρήσεων. Είμαι βεβαία ότι εκπρόσωποι τη Ευρωπόλ θα σα ε, δώσουν ευχαρίστω περισσότερε πληροφορίε για τη δημιουργία αυτού του νέου κέντρου. Στη συνεδρίαση του Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και επίσημα την ενοποιημένη τη έκθεση πεπραγμένων του 2018 ένα έγγραφο που σας ε, είχε στείλει νωρίτερα για διαβούλευση στις αρχές του έτους. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, η κυρία Κατρίν Μπολ έκανε μια συνολική επισκόπηση των στόχων που επιδιώκει η νέα εξωτερική στρατηγική της Ευρωπόλ. Ένα έγγραφο που υπόκειται σε περαιτέρω συζητήσεις και θα ολοκληρωθεί του χρόνου. Το τελευταίο τμήμα της ε, συνεδρίασης ε, περιείχε βρυθείς ε, συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές Ευρωπόλ για το μέλλον και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις δραστηριότητες του οργανισμού. Το πρόγραμμα εργασιών του 2018 απεκάλυψε ότι οι μελλοντικοί δημοσιονομικοί περιορισμοί δημιουργήσαν σε υποβιβασμό σημαντικών σχεδίων και δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ, που αφαιρέθηκαν από το κατάλογο προτεραιοτήτων. Ο κατάλογος αυτών των υπο, υποβαθμισμένων δραστηριοτήτων έγινε τις σημαντικές ανησυχίες των κρατών μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου και έδειξε ότι πραγματικά είναι εύλογες οι ανησυχίες μας. Από αυτή την άποψη, η έλλειψη ε, επενδύσω σε τεχνολογία και εγκληματολογικέ ικανότητε, θα εμποδίσει τον οργανισμό στο μέλλον να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τα, τον ψηφιακό κόσμο. Και επίση, ο αριθμό των συμβασιούχων υπαλλήλων ίσω μειωθεί στο μέλλον και ο οργανισμό ίσω δεν καταφέρει να προσφέρει την επαρκή επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Τέλο, και για να πάμε λίγο πιο μακριά, ο κύριο Σιλίντσα. ε, προσκλήθηκε για να παρουσιάσει τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ε, Δημοσιονομική Αρχή της Ευρωπόλ ε, μέσω επιστολής ε, πριν το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών που έλαβε χώρα σε 6 με 7 Μαΐου 2019. Μάλιστα, αυτή η επιστολή επεστάλλει στον πρόεδρο Ταγιάννη και στην κυρία Κάρμεν Ντάν, την Ρουμάνα Υπουργό Εσωτερικών, στις 4 Ιουνίου του 2017 και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στους συμπροέδρους της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Στη συζήτηση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρθηκαν σημαντικέ σημαντικές πτυχές για τις μελλοντικές δραστηριότητες και την οργάνωση της Ευρωπόλ. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε ώστε να υπερβούμε τις ε, συνεχείς προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Φλωρέα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ευχαρισ... σας ευχαριστούμε που εκπροσωπήσατε στην συνεδρίαση του Μαΐου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ τη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις, θέλει κανείς το λόγο. Ουδής. Καλώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Λίντσα και την κυρία Φλωρέα. Σας είμαστε ευγνώμων, κυρίως, ε, ευγνώμονες κυρία Φλόρα, γιατί ως πρώην συμπρόεδρος μας ενημερώσετε για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ. Και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και θα συνεχίσουμε στις 5 παρατέταρτο. Παρακαλώ να είστε όλοι παρόντες.